sì. Sì, sì, sì, questo. Ok, Allora, <clears throat> buonasera a tutti. Καλησπέρα σα. Να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μα. Να σα θυμίσω ότι θα πρέπει να πάρετε την ηλεκτρονική σας κάρτα για ψηφοφορία, λάβατε την σε διάταξη να σας πω ότι υπάρχει και η μετάδοση στο διαδίκτυο της συνεδρίασης και γνωρίζετε και ποιες είναι οι γλώσσες της συνεδρίασης. Να ξεκινήσω ε, με μια ανακοίνωση. Η συνεδρίαση ΕΚΟΝ 31 Μαρτίου α, ακυρώθηκε. Ας περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία, σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υπονάφτυξης χώρες, εισηγητής ο κύριος Στάες. Θα πρέπει να ψηφίσουμε με βάση τον κατάλογο ψηφοφορίας που έχετε ενώπιόν σας. Αν ε, συμφωνείτε να ξεκινήσουμε αμέσως με την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία υπαριθμών 1. La votazione è chiusa. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 2, άρχεται ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Emendamento 3. Τροπολογία 3, άρχεται ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία περιθμών 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία περιθμών 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία περιθμών 7, αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8, αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Αρχής ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. αρχή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έπειτα ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά. 16 ψήφους υπέρ. Adesso abbiamo il punto... Περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, απαλλαγή 2009, γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή. Πριν να ξεκινήσει η ψηφοφορία, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή που ζήτησε το λόγο. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, παρακαλώ. And... Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και, τους, και τις συναδέλφους που συνέβαλαν στην σύνταξη της λίστας ψηφοφορία. Βέβαια θα ήθελα να είχαν γίνει και άλλες συμβαστικές τροπολογίες, αλλά δοθέντος του χαρακτήρως των τροπολογιών δεν ήταν δυνατόν να γίνουν παραπάνω συμβαστικές τροπολογίες, γιατί είχαν πολλές αποστάσεις μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, έχω τώρα να σας πω τις εξή τροποποιήσεις στην λίστα ψηφοφορίας για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το πρώτο είναι στη σελίδα 4. Η προτινόμενη ψηφοφορία όλες μαζί θα είναι από 44 μέχρι 47 μονάχα, γιατί 43 θέλει το Λαϊκό Κόμμα ξεχωριστά. Υπάρχει και ένα λάθος στη σελίδα 4. Η σύστασή μου για την τροπολογία της κυρίας Ιβάνοβα επί της 66 θα πρέπει να είναι μείον. Στην σελίδα 12 η σύστασή μου για την τροπολογία 172 πάλι πρέπει να γίνει μείον και στην 16 221, τροπολογία 221 έχει αποσυρθεί. Αυτά ήταν τα σχόλια που ήθελα να κάνω και παρακαλώ μπορείτε να προχωρήσετε στην ψηφοφορία. Η κυρία Γκρέσλε, επειδή κυκλοφορεί η φήμη ότι οι τροπολογίες περί staff regulation είναι εκτός αρμοδιότητας της ε, Επιτροπής μας, θέλω να πω για το 171, για τις αποζημιώσεις ταξιδιού που δίνονται άπαξ του έτους στους υπαλλήλους και πρόκειται περί 44.000 υπαλλήλων, δηλαδή 18 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Εγώ λοιπόν βρίσκω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό το στοιχείο αυτό για την Επιτροπή μας και θεωρώ ότι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ασφαλώς θα κινήσουν γη και ουρανό για να κριθεί μη παραδεκτή αυτή η υπόθεση, εγώ βρίσκω ιδιαίτερα περίεργο και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή που επιτρέπει, που θεωρεί παραδεκτές τις τροπολογίες αυτές. Ο κ. Στάις. Πράγματι, λέει ο κ. Χατζημαρκάκης, η νομική υπηρεσία της Ευρωβουλής θεώρησε ότι ορισμένες τροπολογίες που έχουν καταθέσει και η κ. Γκρέσλα και άλλοι για θέματα προσωπικού ότι ίσως είναι μη παραδεκτές εγώ δεν θα συμφωνήσω με την άποψη αυτή. Σας παρακαλώ να ακολουθήσετε την λίστα ψηφοφορίας. Οι τροπολογίες αυτές που θα είναι ίσως δυσχερείς για την νομική υπηρεσία έχουν λάβει ένα μείον ή έχουν χωριστεί με ψηφοφορία κατά τμήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθεί υπόψη το αίτημα της κυρίας Κρέσλε αλλά τα τμήματα εκείνα που ίσως προκαλούν δυσχέρειες στην νομική υπηρεσία να φέρουν το πρόσημα μείον. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ ακολουθήστε την λίστα ψυχοφορίας και έτσι κατά την άποψή μου δεν θα προκύψουν προβλήματα με την νομική υπηρεσία. Και ευχαριστώ και πάλι τις και τους συναδέλφους. Λοιπόν, αν συμφωνείτε, να ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία. Πρόταση απόφασης ε, για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Αν συμφωνείτε, μπορούμε να ψηφίσουμε τι τροπολογίε 1 έως 4 από κοινού. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione Εγκρίνεται. Τροπολογίες 5 και 6 μαζί, άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, καταπίπτουν. Διορθώνει ο πρόεδρος, καταπίπτουν. Ψηφίσουμε τώρα λοιπόν την πρόταση απόφαση για την απόρριψη για τον εκτελεστικό οργανισμό για τα οπτικοακουστικά μέσα. Ζητώ συγγνώμη ο πρόεδρος. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρώτης απόφασης ε, για την Επιτροπή άρχεται η ψηφοφορία. La votazione chiusa. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ. Τώρα ψηφίσουμε την πρόταση απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγή προ τον εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευση οπτικοστικών μέσων και πολιτισμού, ε, τροπολογίε 7 και 8. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione chiusa. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται. Τώρα ψηφίζουμε την... το σύνολο της απόφασης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ και μία αποχή. Ψηφίζουμε την πρόταση απόφασης χορήγησης απελογής προς τον εκτελεστικό Οργανισμό και την Ανταγωνιστικότητα και την Οτομία, σε 9 και 10. La votazione Πέρας ψηφοφορίες εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τώρα την πρώτη απόφαση στο σύνολό τη. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. ψηφοφορία. Εγκρίνονται με 18 ψήφους υπέρ και μία αποχή ψηφίσουμε τώρα την πρόταση απόφασης ε, χορήγησης απαλλαγή στον Εθνικό Οργανισμό Υγεία και τους ε, 11 και 12 άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνονται. Ψηφίσουμε τώρα την πρόταση στο σύνολό τη. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Έγκρινεται με 19 ψήφου υπέρ και μία αποχή. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση απόφαση για την χορήγηση απαλλαγή προ τον Οργανισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Τροπολογίε 13 και 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Έγκρονται. Ψηφίζουμε το, την πρώτη σύνολό τη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 18 ψήφου υπέρ και μία αποχή. Πρόταση απόφαση για τη χωρική απαλλαγή για τον Μιλιστικό Οργανισμό ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, τροπολογία 16. Ε, άρχεται ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρώτη συνολό τη, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά πρόταση απόφαση για την χορήγηση απαλλαγή για τον εκτελεστικό νομισμό έρευνα, ε, τροπολογή 7 και 18, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση στο σύνολό τη, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 19 ψήφου υπέρ και μία αποχή πρόταση απόφασης για το κλείσιμο λογαριασμών. Ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες 19, 20, 21, 22, άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 25. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση στο σύνολό τη. Άρχεται η ψηφοφορία. Κιούσα. Πέρας ψηφοφορίας. Εκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά. Τώρα περνούμε στην ε, ψηφοφορία για την τροπολογία 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε ε, μαζί τις τροπολογίες 44 ε, ε, έως 47. Κιούσα. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 50, άρχεται η ψηφοφορία. Votazione ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 48, αρχή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 55, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 56, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59 σε δύο τμήματα. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 58 διορθώνει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 64, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 65, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66. Ψηφίζουμε τροπολογία 66. Προφορική τροπολογία, άρχεται ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφίζουμε τροπολογία 66. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην προφορική τροπολογία για την τροπολογία 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εκρίνεται. Τροπολογία 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία Για το πρώτο τμήμα, τώρα διευκρινίζω ο ε, ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 69. Άρχη ψηφοφορία για την 69. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71 άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73 άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 72 άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74 άρχεται η ψηφοφορία. Αποκινούμε την 75. 74 και 75 μαζί. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Τροπολογία 77 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνονται. Τροπολογία 76 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Άρχη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Άρχη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Άρχη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 84, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 85, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 89. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ενενήντα πέντε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94. Συγχωρείτε. Ο κύριο Γκάιερ, σύμφωνα με τη λίστα μα, είναι συμβατή η δική μου 92 με την ήδη εγκριθήσα 95. Άρα δεν είναι απαραίτητο ότι εκπίπτει, είναι συμπατή. Έχετε δίκιο. Ψηφίσουμε την 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 96 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 97 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 98, άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 99, άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100, άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 102. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 104 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, αποσύρεται 105. Τροπολογία 106. Ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 107. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία 108, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 109, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Όχι, αποσύρεται. Η 111 αποσύρεται. Η 112. Ψηφίζουμε την 112. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 113. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 114 αρχή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 115 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 116 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 117 αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε αυτή η τροπολογία. Πάμε στην 118 και ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 119. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 123. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 124, 125, 126. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 127. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 128. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 129. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 133. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 134. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 135. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 136. Έρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 138, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 137, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 139, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 140. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 141. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 142 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 143 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 144. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 145. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 146 έρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 147. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 148. Ψηφίζουμε. Το πρώτο τμήμα. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το συμβιβασμό υπαριθμών 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την Τροπολογία 155. Πέρας ψηφοφορίας. Εκρίνεται. Προφορική τροπολογία στην τροπολογία 155. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 156. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 157. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 158. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 159. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 160 έως 163. Άρχεται η ψηφοφορία. Σα... Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 164, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ. Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόεδρε, για την 165 θέλω να υποβάλω μια προφορική τροπολογία εκ μέρους των σοσιαλιστών, παρακαλώ. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο έχουμε ήδη συζητήσει πολλές φορές και έχει να κάνει με το αποδεκτό των τροπολογιών που έχουν να κάνουν με τον ε, κανονισμό προσωπικού. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να ψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες. Οι τροπολογίες αυτές έχουν διακανονιστεί από την Νομική Επιτροπή. Νομίζω ότι η προφορική μας λοιπόν τροπολογία η τροποποίηση αυτή που προτείνουμε θα είχε μέσα το 50 και θα έλεγε τα εξή στα αγγλικά. Σημειώνει ότι η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζεται από την αντίληψη του κόσμου όσον αφορά τη δημόσια δίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι νομοθετικές διαδικασίες εφαρμόζονται και στον κανονισμό προσωπικού και ζητάει από την Επιτροπή να εξυγχρονίσει τον κανονισμό προσωπικού έτσι ώστε ε, να πάψουν απαρχιωμένες ε, διαδικασίες και πιστεύουμε ότι μια σωστή, ε, δια, σωστή εξέλιξη καριέρας, σταδιοδρομίας είναι κάτι θετικό. Αυτά λοιπόν έχω να πω και είναι η προφορική μου τροποποίηση για την 165. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Γκρέσ. Η κυρία Γκρέσ, ευχαριστώ. Αυτή η προφορική τροποποίηση δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Άρα δεν είναι αποδεκτή. Also ich möchte die Antragstellerin noch mal bitten, weil ich habe den Text jetzt mal abgeglichen. So groß sind die Unterschiede. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Πρόκειται για διαφορές απόχρωσης. Αν δεν μπορούμε να την πείσουμε, κρίμα, αλλά θα ήταν μια προσπάθεια. Ο εισηγητής είναι κατά, οπότε προχωρούμε στη ψηφοφορία στις 165. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απροβάτω. 167 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 168 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 170 σε τμήματα. Ε, ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την ε, τροπολογία 171 πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα, τη δεύτερη περίοδο λόγου, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Το τρίτο ουσιαστικά τμήμα, λέει ο πρόεδρος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 172. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 173. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 169. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 174. Άρχεται η ψηφοφορία. Κιούσα. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 175. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 176 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 177 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 178 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 179. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 180. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 181 έως 187. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίες. Εγκρίνονται. Τροπολογία 188. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 189. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 190. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 191. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 192-194 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε τις ψηφοφορίες εγκρίνονται. Τροπολογία 195 ψηφίζουμε. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 196 ψηφίζουμε. Πέρασε ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 197 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 198 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 199 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 200. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 201. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 203. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 204. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 206-209. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 210. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 212. Πρώτο τμήμα. Άρχεται ψυχοφορία. Πέρας ψυχοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας ψυχοφορίας. Απορρίπτεται. Έπειτα ψηφίσουμε μαζί, αν συμφωνείτε, τις τροπολογίες 214 έως 219. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 220. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αποσύρθηκε 221. Τροπολογία 222. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 223. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 224. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 225. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 226. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 227. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 228 έως 244. Άρχεται η ψηφοφορία. Τούσα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 245. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 246. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 247. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 248. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 249. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 250, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 251, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί. Όχι, όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. 273. Ψηφίζουμε την 273. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 274. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 275. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 274. 254, συγγνώμη, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 276. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 277. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 278. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 280. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 279. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 281, πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Ε, πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 282-283 είναι ταυτόσιμες. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται. Τροπολογία 285 και 286 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 287 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 289. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Έγκρινεται. Τροπολογία 290. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 291. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 293. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Παρακαλώ. Την αποσύρω θα ήθελα. Την αποσύρω. 294 Αποσύρεται λοιπόν η τροπολογία 294. Για την 293 τη ψηφίσαμε και την εγκρίναμε. Όχι, την απορρίψαμε, διορθώνει ο Πρόεδρος. Οπότε ψηφίζουμε την 295. Κιούσα. Πέρα ψηφοφορία, εγκρίνεται. Τροπολογία 296. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 297 με προφορική τροπολογία ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. sicuro? Sì. 295 non l'avevamo approvato. Emendamento 299. Τροπολογία 299 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 292. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 300. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τροπολογία 301 ε, και προφορική τροπολογία έρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 302 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 303 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 304 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Αν συμφωνείτε, μαζί ψηφίσουμε τις τροπολογίες 1 έως 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στην Επιτροπή και Κοινωνικών Υποθέσεων, τροπολογίες 1 έω 5 μαζί. 1 έω 5, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνονται. Τροπολογία 6, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 1 έως 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Επιτροπή Μεταφορών. Και εδώ ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 1 έως 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνονται. Επιτροπή Ελευθεριών Δικαιοσύνης Ιστορικών Υποθέσεων. Ε, μαζί ψηφίσουμε την 1 έως 6. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνονται. Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευση. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 2 έως 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνονται. Επιτροπή Περιβάλλοντο Δημοσυγεία και Ασφάλειας Τροφίμων μαζί ψηφίσουμε τροπολογίες 1 έως 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίε. Εγκρίνονται. Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, Τροπολογίε 1 έως 3, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίε. Εγκρίνονται. Και πάλι ψηφίσουμε τώρα τις τροπολογίες 5 έως 7, αρχή ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, τρο, ε, τροπολογίες μαζί 1 έως 7, πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τις τολικές σκέψεις, το υπαριθμών 27. Άρχεται ε, η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 27, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 28, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 29, ψηφίζουμε. Ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 30, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 31, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 32, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 33, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 34. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 35. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Ah, okay. Ritirato αποσύρεται. Διορθώνει ο Πρόεδρος. Αιτιολογική σκέψη 37. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 38. Τροπολογία 38. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Άρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 40 έως 42. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Κιούσα. Πέρας ψηφοφορίας. Έγκρινεται με 21 ψήφους υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Να ευχαριστήσω όλους σας, τον εισηγητή και τους συναδέλφους για ε, τις εργασίες μας. Questo eh, Περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη, που είναι οι ειδικέ εκθέσει του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου στα πλαίσια της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2009 οι ειδικέ εκθέσεις λοιπόν του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου. Ξεκινάμε με την τροπολογία αριθμό 1 παρακαλώ, με 14 μαζί. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τώρα Τη Επιτροπή για τα Δικαιώματα τη Γυναίκα. Τροπολογίε 1 και 2 μαζί. Ψηφίζουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνονται. Τώρα μαζί πάντα τη ίδια επιτροπή 6, 7 και 8. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνονται. Επιτροπή Ανάπτυξης, τροπολογίες 7 μέχρι και 10 μαζί, ψηφίστε. Α, μέχρι και 12. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τώρα ολόκληρο το κείμενο. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 19 υπέρ και μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, 81ο και 10ο, την απαλλαγή του 2009. Ψηφίζουμε την πρόταση απόφαση στο σύνολό τη. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραστη τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ και μία κατά. Η πρόταση απόφαση τώρα για το κλείσμα των λογαριασμών. Το σύνολο της πρότασης. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραστη τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά. Και τώρα περνάμε στις τροπολογίες, το ψήφισμα, τροπολογία αριθμός 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Τέσσερα. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρα στις προφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις προφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ψηφίστε. Πέρα στις προφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Ψηφίστε. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 26. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πρόταση της Επιτροπής Ανάπτυξης τώρα. Μαζί. Μαζί τις τροπολογίες. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί, εφόσον συμφωνείτε. Ψηφίστε παρακαλώ μαζί όλες οι τροπολογίες αυτές. Πέρα στις φοφορίες εγκρινονται εγκρίνονται. Πάντα Επιτροπή Ανάπτυξης μαζί από 18α θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε μέχρι την 1 στην αιτιολογική σκέψη Γ αλλά θέλουμε μείον για την ψηφοφορία κατά τμήματα. <clears throat> θέλουμε, θέλουμε δηλαδή ξεχωριστά. Δεκαοκτώ α. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 18β. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 18Σ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 18Δ. Δέλτα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 18E. Ε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 18F σίγμα Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1 στην αιτιολογική σκέψη Γ. Αρχίζει η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 τώρα στην αιτιολογική σκέψη Δ. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις προφορίες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις προφορίες. Απορρίπτεται. Τώρα First Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 8. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ και μία ψήφος κατά. Και μία αποχή. Όχι, καμία αποχή, καμία αποχή. Συγχαρητήρια. adesso c'è questo, quello dell'altra volta. Adesso abbiamo un... Sì, un attimo, one Volevi intervenire? No? In occasione, eh, per quanto riguarda... ho solo αφορά την πρόταση για την απαλλαγή για το 2009 για την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, Δυστυχώ, σε συζητήσεις που είχαμε στις 22 Μαρτίου, όσον αφορά την απαλλαγή της ΕΟΚΕ, δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση μετά από μια προφορική τροπολογία που προτάθηκε από τον συνάδελφο κύριο Ριβελίνη που δεν έπρεπε να τεθεί σε ψηφοφορία. Αυτή η σύγχυση οδήγησε στο εξή. Δεν ψηφίστηκε η πρόταση απόφασης όπως τροποποιήθηκε. Δυστυχώς αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν, συνέβη όμως. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να ολοκληρώσουμε την διαδικασία ε, απαλλαγής χωρίς να επαναλάβουμε τα πάντα μόνο αυτό το σημείο να ψηφίσουμε την πρόταση απόφασης όπως τροποποιήθηκε. Ο κύριος, η κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ θέλω να εκφράσω την απογοητευσή μου και την έκπληξή μου. Ποτέ δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσα χρόνια. Καταλαβαίνω βέβαια και την απογοήτευση του κύριου Ριβελίνη, ο οποίο ε, μου ζήτησε να κλειστώ μάτια μπροστά σε αυτή την ε, κατάσταση. Και μια που έτσι κι αλλιώ ε, υπάρχει απαλλαγή, θα μπορούσε να ασχοληθώ. Πάντω αυτή τη στιγμή, αν η Όλαφ έχει ανοίξει μια υπόθεση μετά από τόσου μήνε, γιατί πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το μόνο που μπορώ να ζητήσω τη στιγμή τη ψηφοφορία είναι να αναβάλουμε μέχρι την Ολομέλεια, να δούμε πω η Όλαφ έχει να μα πει κάτι καινούριο, να αναβάλουμε μέχρι την Ολομέλεια αυτό το θέμα. Οι συναδελφοί πρέπει να λάβουν υπόψη του ότι βρισκόμαστε και θα μας δικαιώσει σε αυτό η Όλαφ σε μια περίπτωση κακοδιαχείρισης και όσον αφορά τις διαδικασίες, που είναι περίπλοκες και που υπήρξαν και πειθαρχικά ζητήματα και καταδίκη για πληρωμή 7.000 ε, ευρώ που επίση υπάρχουν τέλο πάντων θέματα κακοδιαχείρισης όσον αφορά τον κοινοτικό προπολογισμό. Γι' αυτό και δεδομένου ότι τις προάλλες ε, δεν λέω από πρόθεση, ο κύριος Ριβελίνη πάντως χρησιμοποίησε τρόπους πίσω συνηθίζει να χρησιμοποιήσει το κόμμα του στην Ιταλία, φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση κατάσταση σύγχυσης. Γι' αυτό και σήμερα πρέπει να ε, ψηφίσουμε αυτή την απόφαση όπου είχα μια τροπολογία και το δεύτερο τμήμα που εγώ ε, αιτιολογούσα όλες τις πτυχές αυτής της κακοδιαχείρισης που εντοπίστηκε και που και εσείς ο ίδιος είπατε και στείλαμε το θέμα στην ολάφη η οποία ξεκίνησε έρευνα. Ε, λοιπόν, είχαμε 26 ψήφους υπέρ και μία κατά και καθόλου αποχές από ό,τι θυμάμαι. Τώρα, ψηφίζοντας την απόφαση, αν ψηφίσουμε διαφορετικά, δεν ξέρω, πρέπει να γίνουν κάποιες τεχνικές ε, διορθώσεις. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, το υπόλοιπο ψηφίστηκε με 26 ψήφους υπέρ, μία κατά και καμία αποχή. Φαντάζομαι ότι όλοι με το χέρι στην καρδιά θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ τους συναδέλφους να λάβουν υπόψη τους ότι θέλω να αναβληθεί αυτό το θέμα, αυτή η ψηφοφορία και να περιμένουμε μέχρι να έχουμε περισσότερα στοιχεία από την Όλαφ. Να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία τουλάχιστον μέχρι την Ολομέλεια, για να έχουμε χρόνο να το σκεφτούμε περισσότερο. Η κυρία Γκρέση. Εμείς θα υπερψηφίσουμε την απαλλαγή για ένα απλό λόγο. Στις 13 Μαρτίου 2011 η διαδικασία συνδιαλλαγής μας ανακοινώθηκε από την Όλαφ για, το, για την, για την κοινωνική, επιτροπή, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και είπαμε ότι θέλουμε να γνωρίζουμε για την επόμενη απαλλαγή, μιλάμε τώρα για το 2009, να επανεπεξεργαστούμε το θέμα. Για μένα είναι αδιάφορο εάν θα δοθεί τώρα απαλλαγή ή όχι. Αλλά λόγω των διαδικασιών που έχουν κινηθεί μπορούν να γίνουν και τα δύο. Ακόμα και αν τώρα είμαστε υπέρ τη απαλλαγή, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επεξεργαστούμε τα υπόλοιπα. Και ο επόμενο εισηγητή λοιπόν πρέπει να τα επεξεργαστεί σε βάθο. Φαίνεται ότι πολλούνται έπιπλα στα θεσμικά όργανα σε ιδιωτικούς λογαριασμούς. Πρέπει να εξετάσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι είδους προστασία προσφέρεται στα πρόσωπα που εμπλέκονται στις ε, έρευνες και θα εμφανιστούν πράγματα στη διάρκεια της διαδικασίας της απαλλαγής διότι κάποια στιγμή θα υποχρεωθούμε να μην απαλλάσσουμε πλέον κανένα. Ανησυχώ λίγο διότι κάθε χρόνο ο αριθμός των προσώπων που δεν μπορούμε να απαλλάξουμε μεγαλώνει. Νομίζω λοιπόν ότι για την ώρα μπορούν να γίνουν και τα δύο πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Κύριε Γκρέσλα, δεν αρνούμαστε, αυτό θέλω να επενθυμίσω, δεν αρνούμαστε να το κάνουμε, αναβολή ζητάμε. Να δούμε τι θα πει και ο ΛΑΦ. Μετά από μήνες, ε, γιατί το έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την πρώτη φορά που ζητήσαμε το Σεπτέμβριο να πάει στην όλα αυτό το θέμα η Όλαφ λοιπόν είχε καιρό να το σκεφτεί. Και το μόνο που λέω είναι να αναβάλουμε, δεν λέω να πούμε όχι, λέω να αναβάλουμε αυτό το θέμα. Γιατί αν έρθει Όλαφ και μας πει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ε, θα είναι τα πράγματα τι θα κάνουμε αν υπάρξει πρόβλημα στην Όλαφ. Γι' αυτό ζητάω να αναβληθεί η ψηφοφορία. Δεν λέω να καταψηφίσουμε, να αναβάλουμε λέω. Εσείς κύριε Γκρέσσερ είσαστε υπέρ της αναβολής, όχι. Θέλει κανένας άλλος το λόγο. Η κυρία Γιάλα λοιπόν λέει να αναβληθεί η ψηφοφορία. Η κυρία Γκρέσσερ λέει να ψηφίσουμε σήμερα. Να ψηφίσουμε σήμερα. Τότε ψηφίζουμε την απόφαση απαλλαγής όπως τροποποιήθηκε με την ψηφοφορία της 22ης Μαρτίου 2011. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορία απορρίπτεται με 13 ψήφους κατά, 9 υπέρ και 2 αποχές. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. 11 Απριλίου είναι η επόμενη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στους συγκητές.